ενώ παρακαλούμε τους συναδέλφους της Επιτροπής Προπολογισμών να καθίσουν, παρακαλώ βάλτε την κάρτα σας, να κάνουμε μια δοκιμή, Ζαν Αχτούη παρακαλώ την κάρτα, να προσθέσουμε μια ψήφο από τον Πρόεδρο. Ο, Ζαν δεν έχει την κάρτα του, άρχεται ψηφοφορία για δοκιμή τώρα, έτσι. Γίνεται μια δοκιμή του συστήματος. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία, δοκιμή κάνουμε. Λοιπόν, μπορεί να ολοκληρωθεί η δοκιμή. Ψηφίζουμε τη θέση των αναπληρωτού Γενικού Διευθυντού. Πριν το κάνουμε αυτό, ενημερώσω τις Επιτροπές ότι οι συντονιστές βάσει ομόφωνης αποφάσεως μετά την ακρόαση την περιστατωμένη και οι δύο επιτροπές συνέστησαν στη διάσκεψη των Προέδρων να διοριστεί ο κ. Λάσλο Άντορ σαν ανεξάρτητο μέλος της Διευθύνουσα Επιτροπής του ΕΦΣΥ, οπότε θα προχωρήσουμε στο διορισμό του. Ήταν ομόφωνη η απόφαση. Ε, συγχαρητήρια. Πάμε στην ψηφοφορία για τον κύριο Μόλτερερ, που διορίζεται εκ νέου ο Βίλιαμ Μόρτερ σαν διευθυντής της ΕΦΣΥ. Μυστική ψηφοφορία. Μυστική. Άρχεται η ψηφοφορία. Πιο γρήγορα παρακαλώ. Καλώς. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Πέρας. 44 ψήφοι υπέρ, 2 ψήφοι κατά, 6 αποχές. Οπότε υποψήφιος εγκρίνεται 45. Έχουμε άλλη μία ψήφο. Σας ευχαριστώ. Ψηφίζουμε για την Ιλιάνα Τσανόβα σαν υποδιευθύντρια ξανά εκ νέου διορισμός της, ανανεώνεται ο διορισμός μέσω ψηφτική, ε, συγγνώμη, μυστικής ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. 44 ψήφοι υπέρ, συν μία ψήφος, 3 ψήφοι εναντίον, 5 αποχές, συγχαρητήρια. Και στην Γιάννα Τσενόβα, χειροκροτήματα και για τους δύο και για τον κύριο Άντορ. Πριν ολοκληρωθεί η συνεδρίασή μας, νιοθετήσουμε τα πρακτικά της Δευτέρας Ιουλίου. Τα πρακτικά της τους για τις 2 Ιουλίου δεν υπάρχει αντίρρηση, εγκρίνονται, ολοκληρώνεται αυτή η συνεδρίαση που υπήρξε άκρως αποτελεσματική. Ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Bye bye.